Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, καθίστε. Καλημέρα, συνάδελφοι. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε τη Σύνοδο, να χαιρετήσω και το ακροατήριο. Καλημέρα σας. Άρχεται η σύνοδος. Είναι σημαντική ημέρα σήμερα, όπως ξέρετε. Η ημερήσια διάταξη ορίζει την παρουσίαση του Σώματος των Επιτρόπων και του προγράμματός του από την εκλεγήσα πρόεδρο της Επιτροπής. Οπότε θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ούρσουλα Φοντελέγεν ώστε να κάνει την εισήγηση στην ε, σημερινή συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, Πρόεδρε. The 27th of November. Τον 27 Νοεμβρίου και ακριβώς πριν από 30 χρόνια το ρολόι χτύπησε 12, άρχισαν να ηχούν οι καμπάνες. Οι εργάτες άφησαν τα εργαλεία, τα εργοστάσια, τα ορυχεία και τα μαγαζιά άδειασαν καθώς ε, γέμισαν, πλημμύρισαν ε, οι δρόμοι. Ήταν η ιστορική γενική απεργία στα μέσα της ε, Βελούδινης Επανάστασης που είδε τον κόσμο από το Γκρας, στην Μπρατισλάβα να σειραίει στους δρόμους σε μια ειρηνική ε, έκφραση χαράς. Για μένα αυτές οι δύο ε, αυτή η στιγμή σημαίνει την καρδιά της Ευρώπης. Ε, δεν αφορά μόνο τα κόμματα και την πολιτική, τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις αγορές, τα νομίσματα πάνω από όλα τα άλλα αφορά τον ανθρώπους, του δικές τους προσδοκίες. Πρόκειται για την κοινή προσπάθεια των ανθρώπων, για την ελευθερία, για τις αξίες, για ένα καλύτερο μέλλον απλά. Μια παράθεση από τον σπουδαίο Βάτλαβ Χάβελ, έναν από τους ήρωες του 1989, που για μένα ξεχωρίζει όταν ε, κοιτώ προς το μέλλον. Ε, ε, είπε να δουλεύεις για κάτι επειδή είναι καλό, όχι μόνο επειδή μπορεί και να πετύχει. Διάλεξα αυτή την παράθεση γιατί τα επόμενα πέντε χρόνια η Ένωσή μας θα ξεκινήσει μια μεταμόρφωση που θα αγγίξει κάθε κομμάτι της κοινωνίας μας και της οικονομίας μας. Και αυτό θα το κάνουμε γιατί είναι το σωστό, όχι επειδή θα είναι εύκολο. Κάποιες φορές ξεχνάμε ότι τα μεγαλύτερα μας, τα σπουδαιότερά μας επιτεύγματα προέκυψαν επειδή φανήκαμε τολμηροί. Φανήκαμε τολμηροί για την αναζήτηση της ειρήνης. Όταν δημιουργήσαμε την ενιαία αγορά και το ενιαίο νόμισμα, ήμασταν τολμηροί όταν καλωσορίσαμε ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής μας οικογένειας που ήταν έξω στο κρύο για πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έπρεπε ωστόσο να εστιάσουμε στο εδώ και τώρα, να χειριστούμε τη μία κρίση μετά την άλλη έκτακτη ανάγκη, ε, επίγουσα κατάσταση. Ε, Νομίζω πως έχουμε ωστόσο ε, επανέλθει δρυμύτεροι από αυτές τις δυσκολίες και αυτό χάρη στην ηγετική φυσιογνωμία και τις πεπιθήσεις του προκατόχου μου, του Ζαν Κλοντ Ιούγκερ, ενός σπουδαίου Ευρωπαίου που αφιέρωσε την καρδιά του και τη ζωή του στην Ένωση και το κληροδότημά του μιλά από μόνο του. Ζαν Κλοντ, ευχαριστώ εκ μέρους όλων μας. Κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν από τέσσερις μήνες εσείς ε, μου δώσατε την εμπιστοσύνη σας. Έκτοτε ήρθα σε επαφή με όλες τις πολιτικές ομάδες, όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Μαζί σχηματίσαμε μια ευρωπαϊκή ομάδα εξαιρετική εσείς οι ευρωβουλευτές περάσατε από ακρόαση κάθε έναν από εμά. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας ακούσω και ακριβώ αυτό έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω με την συνοδεία του Μάρκ Σεύκοβιτς και όλων των υπόλοιπων ε, συναδέλφων. Ε, Κάποιες φορές διαφωνήσαμε, κάποιες φορές συμφωνήσαμε, αλλά αυτά είναι η ζωντανή δημοκρατία. Σήμερα εδώ, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, ζητώ τη στήριξή σας για μια νέα αρχή για την Ευρώπη. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, η ομάδα επί της οποίας θα ψηφίσετε σήμερα προέρχεται από διαφορετικούς πολιτισμούς, χώρες, διαφορετικό ιστορικό και πολιτικό και σε αποχρώσεις έχει. Έχουμε δασκάλους, αγρότες, δημάρχους, υπουργούς, γιατρούς, διπλωμάτες, μηχανικούς και επιχειρηματίες. Έχουμε εκείνους που γεννήθηκαν πριν να χτιστεί το τείχος του Βερολίνου και εκείνους που γεννήθηκαν αφού κατερρίφθη εκείνους που έζησαν σε δικτατορίες και εκείνους που ε, βοήθησαν νεαρές δημοκρατίες να μπουν στην Ένωση. Είναι μια ομάδα που σχεδόν έχει ε, τόσες γυναίκες όσο και άνδρους, μόνο μία γυναίκα λιγότερη και φτάσαμε στην ισορροπία των φίλων. Και αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε προοδεύσει, αλλά επίσης ότι πρέπει ακόμα να δουλέψουμε πολύ. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Επιτροπής, επιμένω ότι κάθε μέλος θα έχει ισορροπία στο επιτελείο του. Ισορροπία των φίλων. Και Επίσης θα επιμείνουμε για ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για πρώτη φορά και αυτό θα αλλάξει την όψη της Επιτροπής. Κάθε μέλος της ομάδας μου θα φέρει την δική του προσωπική ιστορία και προοπτική για την Ευρώπη. Θα έχουν τις δικές τους πολιτικές και προτεραιότητες να διαχειριστούν, αλλά όλοι μαζί θα είμαστε μια ομάδα που εργάζεται προς το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Θα είμαστε μια ομάδα που θα συνεργαστεί με, με σας, αυτό το σώμα και τα κρατημέλη για να μπορέσουμε να ορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Αλλά πάνω απ' όλα η Ευρώπη είναι έτοιμη. Το μήνυμά μου είναι στρωθούμε στη δουλειά. Αξιότιμα μέλη, έχουν, πολλοί μιλάνε με αντιπαράθεση στο σημερινό κόσμο και μονομερή προσέγγιση στα θέματα. Αλλά επίσης έχουμε έναν κόσμο που εκατομμύρια άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της διαφθοράς, να απαιτήσουν δημοκρατικές αλλαγές. Ο κόσμος χρειάζεται την ηγεσία μας τώρα περισσότερο από ποτέ. Θα πρέπει να ε, ερχόμαστε επαφή με τον κόσμο σαν υπεύθυνη δύναμη. είμαστε δύναμη για την ειρήνη, για θετική αλλαγή. Να δείξουμε στους εταίρους μας, τα Ηνωμένα Έθνη, ότι μπορούν να βασίζονται σε εμά, θρασπιστέ των πολυμερών συζητήσεων. Να δείξουμε στους φίλους μας τα Δυτικά Βαλκάνια ότι μοιραζόμαστε την ίδια Ήπειρο, την ίδια ιστορία, μοιραζόμαστε τον ίδιο πολιτισμό και θα μοιραστούμε την ίδια μοίρα και πεπρωμένο η πόρτα μας παραμένει ανοιχτή. Επίσης μοιραζόμαστε το ίδιο πεπρωμένο με την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Ναι, έχουμε ζητήματα. Αναμφισβήτητο αυτό. Αλλά οι δεσμοί μας έχουν αντέξει στο χρόνο. Τώρα που μιλάμε, χιλιάδες ερευνητές, φοιτητές, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες εξακολουθούν να, να δημιουργούν μεγάλο αριθμό ε, φιλιών, επιστημονικών προγραμμάτων, μυριάδες ε, προγραμμάτων, ιστοί που διασυνδέονται και δημιουργούν ισχυρό δεσμό, ισχυρότερο από οποιαδήποτε ε, σημείο διαφωνίας. Χώρες από Ανατολή, από Δύση, από Νότο μέχρι το Βορρά χρειάζονται την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πραγματικός εταίρος, το χρειάζονται. Μπορούμε να διαμορφώσουμε καλύτερη παγκόσμια τάξη. Αυτή, αυτός είναι ο στόχος και το πεπρωμένο της Ευρώπης και αυτό θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και χαίρομαι που έχω, μια τέτοια, έχω ένα τέτοιο έμπειρο διπλωμάτη όπως είναι ο Ζιώζεφ Μπορέλ στην ομάδα μου μαζί με την Γιούτερ Πιλάνεν, τον Γιάννη Λένατσικ θα κάνουν ό,τι μπορούν μαζί, θα κάνουν πολύτιμη δουλειά θα επενδύσουμε σε συμμαχίες και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις αξίες μας θα προωθήσουμε και θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης μέσω ανοιχτού και δίκαιου εμπορίου, θα ενισχύσουμε τους εταίρους μας μέσω συνεργασίας, διότι ισχυροί εταίροι κάνουν και την Ευρώπη ισχυρή. Η Ευρωπαϊκή μου Επιτροπή δεν θα φοβηθεί να μιλήσει τη γλώσσα της εμπιστοσύνης, της πεποίθησης, αλλά η ευρωπαϊκή λύση, ο ευρωπαϊκός τρόπος θα ισχύσει. Αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω υπόψη μου και αυτό είναι κάτι που κατεπηγόντω το χρειάζεται η Ευρώπη. Αξιότιμα μέλη, αν υπάρχει ένα ένας τομέας στον οποίο ζητά ο κόσμος να γυθούμε και το έχει ανάγκη, είναι η προστασία του κλίματος. Είναι υπαρξιακό θέμα αυτό για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Πώς να μην είναι υπαρξιακό θέμα. 85% του κόσμου ζει σε ακραία φτώχεια στις 20 χώρες που είναι πλέον ευάλωτες στις ε, αλλαγές του κλίματος. Πώς να μην είναι υπαρξιακό θέμα όταν βλέπουμε τη Βενετία βυθισμένη κάτω από το νερό, τα δάση της Πορτογαλίας να φλέγονται και να χάνει τη σοδιά της κατά το ίμιση η Λιθουανία λόγω ξηρασίας. Αυτό συνέβη πριν, αδιαφυσβήτητα, ποτέ όμως με αυτή τη συχνότητα και ποτέ με αυτή την ένταση και δεν έχουμε ούτε δευτερόλεπτο να χάσουμε πλέον όσον αφορά την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Όσο πιο γρήγορα κινηθεί η Ευρώπη, τόσο μεγαλύτερα τα ωφέλη για τους πολίτες μας, για την ανταγωνιστικότητά μας και για την ευημερία μας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal, είναι κάτι απαραίτητο για μας, για τον πλανήτη μας, για τους λαούς μας, για τις οικονομίες μας. Ο Φρανς Τίμερμανς είναι ο σωστός άνθρωπος για να το κάνει αυτό να συμβεί, να πραγματοποιηθεί. And Και χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που η Κάντε Σίμψον, η Αντίνα Βαλεάν και πολλοί άλλοι θα τον υποστηρίξουν. Η Ευρωπαϊκή αυτή πράσινη συμφωνία, το Green Deal, είναι η νέα μας ε, αναπτυξιακή στρατηγική. Θα περικόψουμε τι εκπομπέ δημιουργώντα θέσεις απασχόλησης. Στο επίκεντρο αυτή της συμφωνίας θα έχουμε βιομηχανική πολιτική που θα δώσει δυνατότητε επιχειρήσει και μεγάλε και μικρέ να καινοτομήσουν και να αναπτύξουν νέε τεχνολογίε ενώ θα δημιουργούν και νέε αγορέ. Θα δημιουργούμε τα παγκόσμια πρότυπα αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσουμε ισότιμου όρου. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να υπηρετούν τους ευρωπαϊκούς λαούς. Θέλουν και προσδοκούν η Ευρώπη να κινηθεί για το περιβάλλον και το κλίμα. Επίσης όμως χρειάζονται καθαρή ενέργεια, ασφαλή ενέργεια, φθηνή ενέργεια. Να έχουν τις δεξιότητες για τις αυριανές θέσεις απασχόλησης, να μπορούν να πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά τους και να συνδέονται από το σπίτι τους και να εργαστούν. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι ανάγκες θα εκπληρωθούν με βιώσιμο τρόπο. Είναι μετάβαση γενεάς για την ουτερότητα του κλίματος μέχρι τα μέσα του αιώνα. Αλλά αυτή η μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιη και συμπεριληπτική. Διαφορετικά δεν θα συμβεί καθόλου. Θα χρειαστεί τεράστια επένδυση για καινοτομία, έρευνα, υποδομές, στέγαση, την κατάρτιση των ανθρώπων θα απαιτήσει και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Για μία ακόμη φορά να πω ότι η Ευρώπη ήδη ηγείται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηματοδότηση του κλίματος θα την λαμβάνει υπόψη ως διαστάση του προπολογισμού αλλά και μέσα στις κεφαλαγορές και σε όλη την αλυσίδα των επενδύσεων σε περιοχές που θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια, θα στηρίξουμε τον κόσμο και τις επιχειρήσεις με στοχευμένη δίκαιη μετάβαση και το σχετικό μηχανισμό θα αφορά διάφορα ταμεία και εργαλεία, θα είναι ζώντια προσέγγιση και θα προσελκύσει ιδιωτικέ επενδύσεις που χρειάζονται για να τα πετύχουμε αυτά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα είναι ένας έμπιστος εταίρος και ιδιαίτερα χαίρομαι ότι η πρόοδος που επετέφθη όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου της σαν μια τράπεζα του κλίματος είναι κάτι προφανές. Θα τονώσει τις επενδύσεις στις ευρωπαϊκές τεχνολογίες και λύσεις που ε, θέλει, χρειάζεται ο κόσμος και τις περιμένει. Αλλά υπάρχουν ε, περισσότερα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Είμαστε περίπου στο 9% από τις παγκόσμιες εκπομπέ, αυτό μας αναλογεί 9%, θα πρέπει ο κόσμος να έρθει μαζί μα. Η φίλιο. αυτό ήδη συμβαίνει από την Κίνα μέχρι τον Καναδά, φτάνοντας μέχρι την Καλιφόρνια. Άλλοι συνεργάζονται μαζί μας για τα δικά του συστήματα εμπορίου ρήπων και ο κ. Χόγκαν θα εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικέ μα εμπορικέ συμφωνίε θα περιέχουν ένα κεφάλαιο για βιώσιμη ανάπτυξη, διότι γνωρίζουμε ότι η αλλαγή του κλίματο μα αφορά όλους και υπάρχουμε καθήκον να δράσουμε και έχουμε και την δύναμη να ηγηθούμε. Κυρίες και κύριοι, η ψηφιοποίηση μας ε, δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουμε πράγματα τα οποία πριν από μία μονογενιά ήταν αδιανόητα. Δηλαδή να επικοινωνούμε με ολόκληρο τον κόσμο, να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, στην έρευνα, στην ε, κινητικότητα, όλα αυτά χωρίς αποκλεισμούς. Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς ε, ψηφιοποίηση. Και η Μαργαρέτε Βεστάγκα είναι εκείνη η οποία θα μας καθοδηγήσει και θα μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. θα αυτοματοποιήσουμε ε, διεργασίες που είναι δύσκολες για τους ανθρώπους. Παραδείγματος χάνει να ανυψώνουν μεγάλα βάρη ή θα μπορέσουμε να αυτοματοποιήσουμε επαναλαμβανόμενες διεργασίες είτε αυτό γίνεται στο εργοστάσιο είτε σε ένα γραφείο. Όμως αυτό έχει και κάτι καλό, δηλαδή θα μας χαρίσει χρόνο χρόνο για εκείνο το οποίο είναι σημαντικό για τους ανθρώπους, είναι εκείνο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και δεν μπορούν να προσφέρουν υπολογιστές. Δηλαδή, ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Παραδείγματο χάρη, έχουμε τα ρομπότ φροντίδας που μπορούν να στρώνουν κρεβάτια και να βοηθούν στην ε, ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Και με τον τρόπο αυτό, το προσωπικό φροντίδας θα έχει και πάλι χρόνο να προσφέρει αυτό που είναι σημαντικό, δηλαδή να συζητά με του τους ασθενείς ε, και να είναι διαθέσιμο για αυτούς. Η ψηφιοποίηση λοιπόν θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικότερα τους φυσικούς πόρους γιατί θα μπορέσουμε να κάνουμε καλή χρήση των υδάτων, της ενέργειας και όλων των αξιόλογων και πολύτιμων πόρων του πλανήτη μας. Ναι, η ψηφιοποίηση είναι εκείνη που θα αλλάξει εκ βάθρων την κοινωνία μας, την οικονομία μας, τη διοίκηση και ήδη συμβαίνει αυτό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτές τις μεγάλες ευκαιρίες και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τους κινδύνους πρέπει να επιφέρουμε την ισορροπία εκεί όπου δεν μπορεί να το πράξει η αγορά. Δηλαδή οφείλουμε να διαφυλάξουμε τόσο την ευρωπαϊκή μας ευμάρεια όσο και τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Πρέπει να ακολουθήσουμε το δικό μας τον ευρωπαϊκό δρόμο και στον χρόνο της ε, ψηφιακής εποχής. Και πώς θα το κάνουμε αυτό. Καταρχήν οφείλουμε να γνωρίζουμε τις τεχνολογίες ε, αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να είμαστε κύριοι των κβαντοεπολογιστών, τη ε, τεχνητή νοημοσύνης, του blockchain, των κριτικών ε, τεχνολογιών των chip. Όμως για να μπορέσουμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά, οφείλουμε να προχωρήσουμε μαζί, να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι είμαστε αποτελεσματικοί. Γι' αυτό α ενώσουμε τους πόρους, α ενώσουμε τα χρήματά μας, την έρευνά μας, τη γνώση μα και όλα αυτά να τα μεταφέρουμε στην πράξη. Ήδη το καταφέραμε μια φορά στον σούπερ υπολογιστή. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ε, πρόκειται να ε, κατασκευάσει έναν από τους μεγαλύτερους και αποδοτικότερους υπολογιστές. Εξαιρετικό αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα αυτόν τον υπολογιστή να τον κατασκευάσουμε, τουλάχιστον κατά την επόμενη γενιά, μόνοι μας ως Ευρωπαίοι. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Η Ευρώπη έχει τους επιστήμονες, έχει όλη εκείνη τη τεχνογνωσία που της χρειάζεται για να είναι ανταγωνιστική και γι' αυτό ας μην το υποτιμούμε. Ας μην το υποτιμούμε και ας μην το δεχόμαστε να μας υποτιμούν ούτε οι άλλοι, αλλά ούτε και μόνοι μας τον εαυτό μας. Η καινοτομία χρειάζεται ευφύης ανθρώπους, αλλά χρειάζεται και διαφοροποίηση. Χρειάζεται ένα περιθώριο για να μπορεί να σκέπτεται. Και όλα αυτά τα έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι θέλουν εδώ να ζουν, εδώ εδώ να κάνουν έρευνα, εδώ να διαμορφώνουν το μέλλον τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν την υποδομή να έχουμε κοινά ε, πρότυπα και προδιαγραφές, ε, δίκτυα ε, cloud τα οποία θα μπορούμε να παραδώσουμε και στην επόμενη γενιά. Ε, η πρώτη ύλη της ψηφιοποίησης είναι τα δεδομένα. Με κάθε κλικ το οποίο κάνουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, με κάθε τέτοιο χτύπημα, τροφοδοτούμε τους αλγόριθμους, κατά κύριο λόγο όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι οποίοι βέβαια με τη σειρά τους επηρεάζουν εμάς, επηρεάζουν τις πράξεις μας. Και αυτό δεν είναι καλό. Για το λόγο αυτό, όπως ακριβώς το πράξαμε και με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, δηλαδή εκεί θέσαμε το πλαίσιο για τον κόσμο και αυτό μπορούσε να το κάνει μόνο η Ευρώπη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πρέπει να το επιτύχουμε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί εμείς ε, στην Ευρώπη ε, σκεπτόμεθα κυρίως τον άνθρωπο, όχι την αγορά, όχι τα χρήματα, όχι το κράτος. Κυρίως στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Και το σημαντικότερο είναι να αναχαιτήσουμε μάλλον εμείς να θέσουμε τους κανόνες, το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, όχι να αναχαιτήσουμε τα δεδομένα. Γιατί για μας, για τους Ευρωπαίους, η προστασία της ε, ψηφιακής ταυτότητας είναι η πρώτη και το πρώτο και κυρίαρχο μέλημά μας. Για μας αυτό είναι το σημαντικότερο. Και παράλληλα επιθυμούμε την κοινοτομία. Σήμερα το 85% όλων των δεδομένων που δεν έχουν σχέση με άτομα, το 85% αυτών των δεδομένων δεν χρησιμοποιούνται ούτε μία φορά. Αποθηκεύονται αυτοματοποιημένα βέβαια, αλλά δεν χρησιμοποιούνται ούτε μία και μόνο φορά. Και αυτό αποτελεί μία τεράστια διασπάθηση, γιατί σε αυτά τα δεδομένα υποκρύπτονται ε, γνωστικά στοιχεία, γνώσεις που πρέπει να τις χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Άρα δηλαδή πρέπει να καθορίσουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και ε, δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν ικανότερο από τον Thierry Breton ο οποίος θα καθορίσει μια στρατηγική για τη χρήση των δεδομένων. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα ε, της ε, κυβερνοασφάλειας που είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, η άλλη πλευρά της ψηφιοποίησης. Άρα και αυτό για μας είναι προτεραιότητα. Για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρειαζόμαστε ύψιστη ασφάλεια, μια ευρωπαϊκή πορεία και ως εκ τούτου οφείλουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για τους κινδύνους need to know, need to share. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια κοινή πλατφόρμα, κατά κάποιον τρόπο αν θέλετε, μια διευρυμένη υπηρεσία για την κυβερνοσφάλεια. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να μπούμε στην δικτυωμένη οικονομία, να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τους κινδύνους και όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα επιτύχουμε μόνο εφόσον προχωράμε όλοι μαζί ενωμένοι μόνο εφόσον βασιζόμεθα στις ευρωπαϊκές μας αξίες. Και είμαι αισιόδοξη ότι η Ευρώπη και στην εποχή της ψηφιοποίησης θα είναι πρωτοπόρα, θα καθορίζει τον δρόμο. Αυτό μπορεί να το επιτύχει η Ευρώπη. Αξιότιμα μέλη, μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλά πράγματα η Ευρώπη. Είμαστε υπερδύναμοι στο εμπόριο στον κόσμο. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο στην εξαγωγή μεταποιημένων βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών. Είμαστε η μεγαλύτερη πηγή και προορισμός ε, των, ξένων ε, άμεσων επενδύσεων στον κόσμο. Οι βιομηχανίε μας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική και παράγει το 1 τρίτο των δορυφόρων στον κόσμο. Και οι εταιρείε μας είναι στην αιχμή έχοντας 40% ε, των αδειών ευαισθητεχνία όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και τη σχετική τεχνολογία. Θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μεταμορφωτική δύναμη τη ε, διτή μετάβαση για το κλίμα και για την ψηφιακή τεχνολογία. Ενισχύσουμε την βιομηχανική μα βάση και τη δυνατότητά μα για καινοτομία. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω των επενδύσεων. Και αξιότιμα μέλη, πρέπει να αυξήσουμε την κλίμακα για χρόνια επενδύουμε λιγότερα στην καινοτομία από ό,τι οι ανταγωνιστέ μα. Αυτό είναι τεράστιο μειονέκτημα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά μα και τη δυνατότητά μα να ηγηθούμε σε αυτή τη μετάβαση και τη μεταμόρφωση. Γι' αυτό δεν πρέπει να θεωρήσουμε το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σαν μια απλή λογιστική άσκηση. Πριν από 7 χρόνια ο κόσμος δεν έχει καμία ομοιότητα με τον κόσμο όπως θα είναι σε 7 χρόνια. Ο κόσμος θα πρέπει να ξυγχρονιστεί σε σημαντικό βαθμό. Σε αυτόν τον τομέα δεν μπορώ μόνο να βασιστώ στην εμπειρία και τις δεξιότητες του Ιωάννης Χάν, αλλά επίσης και σε αυτό το κοινοβούλιο. Αλλά οι δημόσιοι προπολογισμοί έχουν τα όρια τους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η επένδυση μπορεί, μπορεί να ρεύσει εκεί που χρειάζεται συμπληρώνοντα την Ένωση των Κεφαλαγορών. Έτσι θα βελτιώσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, Έτσι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να αντιμετωπίσουν του αναγκαίου κινδύνους. Το ίδιο ισχύει για την Τραπεζική Ένωση. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί, ούτω ώστε το χρηματοπιστωτικό μα σύστημα να γίνει ισχυρότερο και ανθεκτικότερο. Έχω αναθέσει αυτό το καθήκον στον Βάλτι Ντομπρόφσκη. Είναι ο σωστό άνθρωπο για αυτή τη σωστή δουλειά. θα εξασφαλίσει ότι η οικονομία μας θα λειτουργήσει για τον κόσμο. Ποιοτικέ τη απασχόληση, ευκαιρίε, δίκαιε συνθήκε εργασία και να συμπεριλαμβάνονται όλοι. Γνωρίζει ότι χρειαζόμαστε ορθή δημοσιονομική προσέγγιση για βιώσιμη ανάπτυξη και θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητά μας και την βιωσιμότητά μας. Πάνε χέρι με χέρι αυτά. Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ανταγωνιστική βιωσιμότητα πάντα ήταν στο επίκεντρο, στην καρδιά της οικονομίας μας, της αγοράς, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Απλώς την ονομάζαμε διαφορετικά. Τις οικογενειακές επιχειρήσεις σκεφτείτε σε όλη την ένωσή μας. Δεν δημιουργήθηκαν μόνο σε αξία μετοχών ή τις νέες αμοιβέ των στελεχών, βασίστηκαν για να ε, διαρκέσουν και να πάνε από γενιά σε γενιά και να δώσουν ένα δίκαιο βίο στους ε, εργαζομένους. Με πάθος δημιουργήθηκαν για ποιότητα, για παράδοση, για καινοτομία. Αυτά που φτιάχνουμε σήμερα ίσως να έχουν αλλάξει, αλλά θα πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου την ανταγωνιστική μας βιωσιμότητα. Αγαπητοί μου φίλοι εδώ, σε αυτό το σώμα, σε αυτό το πνεύμα, κάθε κράτος μέλος δεσμεύτηκε να πετύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Και σε αυτό το πνεύμα ο Πάολο Τζεντιλόνι θα υποπτεύει την υλοποίηση αυτών των στόχων. Πιστεύεις σε αυτούς και εγώ πιστεύω σε αυτόν. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει ανακάμψει μετά από μια μεγαλύτερη, οικονομική και χρηματοσυντική κρίση μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται. Όμως βλέπουμε νέφη στον ορίζοντα να διαμορφώνονται και θα πρέπει να ετοιμάζεται η Ευρώπη για αυτά που έρχονται. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτό που μας ισχυροποιεί, την ενιαία αγορά το ενίο νόμισμα. Και έγκυκε η ώρα να ολοκληρώσουμε την οικονομική και νομισματική μας ένωση, να πετύχουμε ανάπτυξη θέση απασχόλησης, αυξάνοντας μακροοικονομική αντοχή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία που επιτρέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για να δώσουμε το χρόνο και το χώρο για να αναπτυχθούν οι οικονομίες μας. Ταυτοχρόνως θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη με στοχευμένες επενδύσεις, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο άτομο να ηγηθεί αυτού του έργου από την Ελίζα Φερέιρα. Αξιότιμα μέλη. Τον περασμένο μήνα 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ε, μέσα σε ένα φορτηγό. Οι άνθρωποι αυτοί διέσχισαν τουλάχιστον τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι λοιπόν τραγωδία το ότι μία μητέρα στο Βιετνάμ παίρνει ένα μήνυμα από την κόρη της ε, στην Ευρώπη ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, ότι δεν έχει περιθώριο για να αναπνεύσει. Για αυτούς λοιπόν τους 39 ανθρώπους, για τις μητέρες, τους πατέρες, τους φίλους, όλοι συμφωνούμε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί ποτέ. Οι άνθρωποι περιμένουν από την Ευρώπη να βρει ε, κάποια λύση για την πρόκληση της μετανάστευσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει διχάσει. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε μπροστά. Χρειαζόμαστε λύσεις ε, που θα είναι ικανοποιητικές για όλους. Και ε, αυτό το ανέθεσα στους κυρίους Χινά και Γιώχανσεν που έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, διαφορετικές προοπτικές, αλλά θα αποτελούν ένα μοναδικό ντουέτο. Αξιότιμα μέλη. Ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές. Η Ευρώπη πάντα θα προσφέρει καταφύγιο σε εκείνους οι οποίοι χρειάζονται την διεθνή προστασία. Και είναι λοιπόν προς το συμφέρον μας να παραμείνουν όλοι αυτοί ενταγμένοι στις κοινωνίες μας, αλλά οφείλουμε επίσης ε, να διασφαλίσουμε ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν, θα πρέπει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. πρέπει να σπάσει πια αυτό το βίο εμπορικό μοντέλο των διακινητών. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις αξίες μας που είναι η αλληλεγγύη και η ανάληψη ευθυνών. Οφείλουμε να ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε ένα εύρυθμα λειτουργούν Schengen, σύστημα Schengen Οφείλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες στις χώρες προέλευσης των μεταναστών, να τους προσφέρουμε εκεί ευκαιρίες. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο, αλλά ας μην ξεχνάμε αυτά που είπε ο Χάβελ, που είπε ότι ε, πρέπει κανείς ε, να πράττει και να πράττει το καλό. η μετανάστευση δεν θα εξαφανιστεί, θα παραμείνει. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μια Ευρώπη που είναι τόσο μα τόσο υπερήφανη για τις αξίες της και τόσο υπερήφανη για το κράτος της δικαίου, μια τέτοια Ευρώπη πρέπει να βρει μια απάντηση που θα είναι και ανθρώπινη και αποτελεσματική. Πρέπει να μπορέσουμε να το καταφέρουμε ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς και ο κύριος Γιώχανσεν θα είναι επίσης αρμόδιοι για την ενίσχυση της εσωτερικής μας ασφάλειας. Θα διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή του νόμου θα είναι αποτελεσματική απέναντι στις νέες προκλήσεις και επίσης θα διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη θα έχει την καλύτερη δυνατή εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Αξιότιμοι βουλευτές, όταν εγώ ήμουν νεαρά, μικρό κορίτσι και ζούσα στις Βρυξέλλες, η μικρή μου αδελφή πέθανε σε ηλικία 11 ετών από την όσο του καρκίνου. Και θυμάμαι την ε, απελπισία των γονέων μου, αλλά και των ιατρών της ιατρικής ε, ομάδας που την φρόντισε με τόσο μεγάλη στοργή όλοι μας έχουν να διηγηθούν κάποια ιστορία, είτε στην οικογένειά τους, είτε γνωρίζουν κάποιον που έχει προσβληθεί από καρκίνο. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη διάγνωση και καλύτερες ε, θεραπείες. Η Ευρώπη θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος στον αγώνα κατά του καρκίνου, στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Την επόμενη χρονιά η κυρία Κυριακίδη θα παρουσιάσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου και είναι το σωστό άτομο έτσι ώστε να μπορέσουμε στην Ευρώπη να περιορίσουμε τον πόνο που προκαλεί αυτή η ασθένεια. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να μεριμνά για τα θέματα που αφορούν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το μέλλον των παιδιών τους, για το μέλλον της κοινωνίας. Ο πολιτισμός και η παιδεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ιστορία μας, αλλά και με το μέλλον μας. Και αυτό μας καθιστά μοναδικούς. Η ψυχή μας, ο πολιτισμός μας, μας ε, η πολυμορφία, η κληρονομιά μας, η Μαρία Γκαμπριέλ είναι εκείνη που θα τα φροντίσει όλα αυτά. Είναι σε καλά χέρια αυτά που προανέφερα και με χαρά ανακοινώνω ότι το χαρτοφυλάκιό της θα μετονομαστεί σε Επίτροπο για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και την Νεολαία. Οι άνθρωποι ε, θέλουν δικαιοσύνη και ισότητα με κάθε απόχρωση αυτών των όρων. Γι' αυτό και επέλεξα τον Νίκολα Σμιτ, ο οποίο θα αναλάβει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την ε, καταπολέμηση της φτώχειας ήδη από την παιδική ηλικία. Θα ορίσει ένα πλαίσιο έτσι ώστε κάθε εργαζόμενο στην Ένωσή μας να έχει ένα δίκαιο κατώτατο μισθό. και η Χέλενα Ντάλι θα είναι σκαπανέας για να σπάσουμε τους φραγμούς, οι φραγμοί που δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να γνωρίζουν ποιοι είναι, γιατί πρέπει να αγαπούν και σε τι πρέπει να πιστεύουν αυτοί οι φραγμοί πρέπει επιτέλου να εξαφανιστούν. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματά του, τι αξίε του, τι ελευθερίε του. Το κράτο δικαίου είναι τα θεμέλια μα και αυτό ποτέ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι το κράτο δικαίου γίνεται σεβαστό, κάθε χώρα φροντίζει για το κράτο δικαίου. Βεβαίω και καλλιεργούμε το διάλογο και την πρόληψη, αλλά και ποτέ δεν διστάζουμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Χρειαζόμαστε εμπειρία στράτευση και η Βέρα Γιούροβα και ο Didier Reinders είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να εξασφαλίσουν όλα αυτά. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον αέρα που αναπνέουν, το νερό που πίνουν, τα τρόφιμα που καταναλώνουν και την φύση που τους περιβάλλει. Ε, νομίζω όλοι μας πρέπει να είμαστε ευτυχείς για το ότι ο Βιρτζίνιου Σιντσεβίτσιους ε, θα ε, προσπαθήσει να διασφαλίσει τη βιοπικιλότητα στους ε, ωκεανούς και στην Αλία. Και έχουμε και τον Γιάννους Βοτσεκόψκι, ο οποίος θα εξασφαλίσει ότι οι αγρότες μας θα μπορούν επίσης να προοδεύουν καθώς θα προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα έχουμε τη μετάβαση ε, στο θέμα του κλίματος και στην ψηφιοποίηση. Και αυτό το δίδυμο θα φέρει αλλαγές σε όλους μας, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Η γεωργία θα παραμείνει ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας και του μέλλοντός μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν την βιώσιμη γεωργία, την απαραίτητη στρατηγική, ε, από το νερό γεωργό μέχρι και το εργοστάσιο. Ε, οι εισαγωγέ από τις τρίτες χώρες οφείλουν να είναι συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον. Εξάλλου, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να έχουν και λέγην στο μέλλον τους. Βλέπουμε οι ευρωπαϊκές εκλογές ε, αυτή τη φορά είχαν τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση που υπήρξε ποτέ, αλλά η δημοκρατική συμμετοχή δεν σταματά την ημέρα των εκλογών. Εμείς θα κινητοποιήσουμε τα καλύτερα μυαλά της Ευρώπης ε, σε επίπεδο θεσμών, στην καθημερινότητα, ε, να συμμετέχουν όλοι αυτοί στη συνδιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, όπου δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί, θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι θεσμοί, όλοι οι πολίτες και το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει καθοδηγητικό ρόλο. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η Ντουμπράφκα Σούιτσα ε, θα εργαστεί για να καταστεί όλο αυτό επιτυχία. Αξιότιμα μέλη. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ένα μέλος της οικογένειάς μας ε, προτίθεται να εγκαταλείψει την Ένωση. Μια μεγάλη πλειοψηφία των ε, βουλευτών ε, μοιάζουν να είναι ικανοποιημένοι με το ότι ένα πολύ μικρό κομμάτι δεν θα είναι πια σε θέση να χειροκροτά εκεί που δεν πρέπει. Και νομίζω εγώ ποτέ δεν απέκρυψα το γεγονός ότι εγώ πάντα θα είμαι remainer θα είμαι ο παντός της πολιτικής της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια θα σεβαστούμε την απόφαση που έλαβαν οι Βρετανοί πολίτες. Θα συνεργαστούμε για να ζητήσουμε λύσεις απέναντι στις κοινέ προκλήσεις, κυρίως όσον αφορά θέματα ασφάλειας. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές. Ό,τι και αν φέρει το μέλλον, η δεσμή, η φιλία που ενώνει τους λαούς μας, αυτά είναι άρρηκτα στοιχεία συνδεμένα μεταξύ τους και ποτέ δεν θα πάψουν να υπάρχουν. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, σε 30 χρόνια άλλοι εδώ, σε τον ίδιο χώρο, θα ε, κρίνουν τις ε, ε, δικές μας ενέργειες, όπως το έκανα και εγώ στις αρχές της ομιλίας μου τι θα πούν τότε. Αυτό εξαρτάται από το τι εμείς ε, θα κάνουμε από κοινού. Εάν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, η Ευρώπη του 2050 θα είναι η πρώτη ήπειρος του κόσμου που θα είναι ουδέτερη σε άνθρακα και θα είναι και μια ισχύς, μια δύναμη πρώτης τάξης στο ψηφιακό κόσμο. Επίσης, ε, στην οικονομία θα έχει εξασφαλίσει την ισορροπία ανάμεσα την αγορά και κοινωνικά ζητήματα και επίσης θα είναι πρωταγωνιστή στην επίλυση των μεγάλων ε, προβλημάτων του κόσμου. Ο δρόμος είναι δύσκολος, το έργο δεν είναι εύκολο, αλλά μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ας εμπνευστούμε από αυτό το αισιόδοξο πνεύμα ε, που ίσχυσε πριν από 30 χρόνια που οδήγησε στην πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Για να επανέλθω στο Βάσλαβ Χάβελ υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι που ε, δεσμεύονται γιατί είναι αυτός ο σωστό δρόμο. Υπάρχουν εκείνοι που επενδύουν για να ενισχύσουν την ε, κοινωνία τους, ε, την κοινότητά τους. Υπάρχουν εκείνοι που ε, προσφέρονται για να φροντίσουν ηλικιωμένου, για να καθαρίσουν ένα πάρκο. Εκείνοι που αλλάζουν τη το ζωή τους, τον τρόπο ζωής τους για να προστατέψουν το κλίμα. Άνθρωποι που θέλουν να σημάνουν τη διαφορά. Και εμεί εσύ, και εμεί εδώ, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή και εμείς οφείλουμε να ε, σημάνουμε τη διαφορά. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα έφτιαξα την ομάδα μου και σε αυτό το πνεύμα βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιόν σας για να ζητήσω την εμπιστοσύνη σας. Ας στρωθούμε λοιπόν στη δουλειά ώστε να μπορέσουμε να λέμε σε 30 χρόνια «Ζήτω η Ευρώπη». Ζήτω η Ευρώπη σε όλες τις γλώσσες.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 την Πρόεδρο Βάντερ Λάιν. Χαιρετίζω και εγώ το Συμβούλιο και όλους τους παρόντες επιτρόπους. Ξεκινάμε τη συζήτηση ακούγοντας τους ε, Προέδρους των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει ο Μάνφρετ Βέμπερ. Ορίστε. Λοιπόν, προτεραιότητες αφής και ισορροπία. Αυτά μας είπε η Ρουσούλα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν πολύ σημαντικέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξετάσαμε όλου του υποψηφίου που πρότειναν τα κράτη-μέλη και να δούμε αν είναι έτοιμοι για τη δουλειά. Δεν ήταν όλοι έτοιμοι για τη δουλειά του, αλλά τελικά τώρα έχουμε επιτρόπου μπροστά μα και η ανάλογη, η, αρμόδια επιτροπή έδωσε το πράσινο φω. Το ΕΛΚ εργάστηκε άκνο και εργάστηκε με διαφάνεια στην όλη διαδικασία τελευταίες εβδομάδες και μήνες ήταν ε, δύσκολη η περίοδος για σας, αλλά εσείς τελικά υπήρξατε επιτυχέστατοι, εργαστήκατε ε, άοκνα και μας παρουσιάσατε σήμερα το νέο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ομάδα που θα ηγηθεί για την Ευρώπη. Μαζί πετύχαμε αποτελέσματα και σήμερα ελπίζουμε την πλήρη υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Μπορούμε επίσης να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ε, ισχυρή δημοκρατική νομιμότητα. Ένα από τα βασικά τη ομάδα σα είναι η καλύτερη ισορροπία των φύλων, η βελτίωση τη ισότητα των φύλων. Έχουμε περισσότερε γυναίκε επιτρόπου από ποτέ. Και με υπερηφάνεια λέγω σαν μέρο του ΕΛΚ, σαν πολιτικό ο του ΕΛΚ, ότι πλευρά ΕΛΚ έχουμε 50% γυναίκες. Εμείς πετύχαμε το στόχο μας να έχουμε 50% ισορροπία. Άλλοι ακόμα πρέπει να εξεργαστούν το θέμα και σαν ΕΛΚ έχουμε την πρώτη πρόεδρο Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμά δεν είναι μόνο ευχολόγια και λόγια, εμείς τελικά πραγματοποιούμε την ισορροπία των φίλων. Και έχουμε ένα καλό μείγμα Έχουμε έμπειρου συναδέλφου όπω τον Hans Χάν, τον Φιλ Χόγκαν, Βάλι Ντομπρόφσκη και τη Μαρία Γκαμπριέλ. Έχουμε νέου επιτρόπου όπω τη Στέλλα Κυριακίδη, τον Μαργαρίτη Σχενιά και τον ε, Όλιβερ Βαχίλη και έχουμε δύο συναδέλφους που υπηρέτησαν επί σειρά ετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αντίνα Βαλιάν και Ντουμπράφκα Σουίτσια. Από την ομάδα μας σαν ΕΛΚ έχουμε ένα καλό μείγμα και βασιζόμαστε στη συνεισφορά τους. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ομάδα μου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 40 εκατομμύρια ψήφους πήρε στις τελευταίες ευρωεκλογές και τώρα έχουμε την ευθύνη να δώσουμε αποτελέσματα. Αυτό που οι ψηφοφόροι μας ζήτησαν να κάνουμε σαν μεγαλύτερο κόμμα στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σαν ομάδα θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Το 2024 θα έχουμε εφαρμόσει φιλόδοξο και έξυπνο πρόγραμμα για το κλίμα βάσει καινοτομίας χωρίς να επιτεθούμε κατά των γεωργών και να μην πολιτοκολογούμε κατά της βιομηχανίας. Το 2024 θα έχουμε πετύχει το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα μεγάλο σχέδιο κατά του καρκίνου θα έχουμε πετύχει το 2024 να έχουμε δημιουργήσει 5 εκατομμύρια νέε θέσει απασχόληση και θα πρέπει να σταματήσουμε τη φυγή εγκεφάλων από την Ανατολή, και από την Ανατολή προς Δύση. Το 2024 έχουμε συμφωνήσει για περαιτέρω εμπορικέ συμφωνίε. Όταν ο Τραμπ χτίζει τείχου εμπορικού, εμεί, αν Ευρωπαίοι, θα πρέπει να οικοδομήσουμε γέφυρε εμπορίου. Το 2024 θα έχουμε μεταμορφώσει την Ευρώπη. Η Ευρωπόλ θα έχει γίνει Ευρωπαϊκή FBI θα κινηθεί κατά του οργανωμένου εγκλήματο και τη μαφία. Το 2024 θα έχουμε καθορίσει τα τελικά σύνορα της Ευρώπης. Η Τουρκία είναι ισχυρός εταίρος, αλλά η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το 2024 θα έχουμε δημιουργήσει ευρωπαϊκή μεθοριοφιλιακή και ακτοφυλακή με τουλάχιστον 10.000 ε, υπευθύνου που θα προστατεύουν τα σύνορα και δεν θα αποφασίζουν άλλοι για μας. Αυτό εννοούμε όταν λέμε για αποτελέσματα, γιατί το, το ΕΛΚ σήμερα θα υπερψηφίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α ξεκινήσουμε τώρα, ούτω ώστε να ανταποκριθούμε στι υποσχέσει μα, υλοποιήσουμε τι υποσχέσει. Φιλόδοξα προγράμματα είναι σημαντικά, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά τα επόμενα χρόνια υπάρχουν πολλά ακόμα διακυβεύματα. Αισθανόμαστε ότι οι κοινωνίε μα ε, διαλύονται. Το ευρωπαϊκό κοινό συνέστημα δέχεται συνεχώ ε, επιθέσει διότι υπάρχει διχασμό. Υπάρχουν αυτοί που αισθάνονται ότι απειλούνται την παγκοσμιοποίηση και εκείνοι που αλαμβάνουν τι νέε ευκαιρίε αυτό που κάνει την Ευρώπη η μοναδική ε, κινδυνεύει. Ένα συνέστημα του ανήκειν απαιτείται πολύ. Ταυτότητα χρειάζεται πάρα πολύ. Όλοι μας γνωρίζουμε πώς να περιγράψουμε την εθνική μας ταυτότητα μέσω ιστορίας, μέσω επιτευμάτων του πολιτισμού μας. Αλλά σαν Ευρωπαίοι μπορούμε να περιγράψουμε τους εαυτούς μας, τον τρόπο ζωής μας, ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ακόμα και στοχότερες χώρες της Ευρώπης Έχουμε σύστημα υγείας που βασίζεται σε αλληλεγγύη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα συζητούν το Obamacare. Όλη, σε όλη την Ευρώπη έχουμε απαγόρευση θανατικής ποινή. Αυτό δεν ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ισότιμη αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών και ο ευρωπαϊκό τρόπος ζωής μετά την πτώση του Βερολίνου εδώ και 30 ε, χρόνια, ανεξιθρησκεία, ελευθεροτυπία, ελευθερία του λόγου, ε, ο κινέζικο πολιτισμό με ενδιαφέρει πολύ. Αν θέλω να ζήσω τον κινέζικο τρόπο ζωή, οι Αμερικάνοι πάντα θα είναι ο στενότερο εταίρο Ευρώπη. Δεν θέλω όμω να ζήσω με τον αμερικανικό τρόπο ζωή. Εγώ προτιμώ τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Πάντα θα προστατεύουμε, θα προωθούμε και θα εγγυόμεθα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Μ' αρέσει να είμαι Ευρωπαίο. Τα επόμενα πέντε χρόνια θα αποφασίσουμε κατά πόσο η Ευρώπη θα διατηρήσει την ψυχή τη και την καρδιά τη ή αν θα παραμεριστεί και θα κινηθεί σε έναν πιο βίο τρόπο. Ε, κόσμο, συγγνώμη. Θα συνεργαστεί το ΕΛΚ με όλε τι δημοκρατικέ ομάδε του Κοινοβουλίου για μια καλύτερη Ευρώπη. Το ΕΛΚ έχει αποδείξει ότι είναι, βασίζεται στον Άντε Αντενάου, στο Σούμαν, τον Χέλμουντ Κόλ και τον Γκάσπαρη. Βασιστήκαμε πάνω σε αυτού και κινηθήκαμε για ενωμένη Ευρώπη. Βασίζεται ο κόσμο σε εμά. Α αρχίσουμε τώρα να δίνουμε αποτελέσματα. Σα ευχαριστούμε, Πρόεδρε Βέμπερ. Η πρόεδρος Γκαρσία Πέρες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Βαντερ τον Ιούλιο σας δώσαμε καταρχάς ε, την, την εμπιστοσύνη μας, παρότι δεν ήσασταν υποψη, δική μας υποψήφια, γιατί υποσχεθήκατε να περιλάβετε στο πρόγραμμά σας κάποιες προτεραιότητες που για μας είναι θεμελιώδεις. Είπατε ότι η οικολογική μετάβαση θα είναι το πρώτο θέμα της επόμενης αιτίας και επιπλέον υποσχεθήκατε να το κάνετε με δίκαιο τρόπο χωρίς να μείνει κανένας πίσω. Θα θέλαμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά χρειάζεται να έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν θα μας ε, ε, εξαπατήσει οι σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, την τελευταία μας ψήφο, ε, την τελική μας ψήφο μάλλον, την εξαρτάμε από το γεγονός ότι αυτός ο σπουδαίος στόχος, ε, οικονομική και κοινωνική και περιβαλλοντική μετάβαση, να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που θα βελτιώσει τη ζωή των λαών μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και γι' αυτό μας έχουν εκλέξει. Για να, ε, για να ε, εγγυηθούμε λοιπόν τι αρμοδιότητε και τις ικανότητες του κάθε επιτρόπου, ε, εμείς δουλέψαμε με απαιτητικό τρόπο κατά τη διάρκεια των ακροάσεων των 26 επιτρόπων που θα αποτελέσουν το μελλοντικό σας ε, συλλογικό όργανο, γιατί σε αυτό δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Δεν μπορούμε να αποτύχουμε απέναντι στους νέους που κάθε Παρασκευή διαδηλώνουν για να μας πούν ότι ανησυχούν για το μέλλον τους. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε, γιατί μπορέσατε να δώσετε, να μας προσφέρετε την πιο ισότιμη όσον αφορά το φύλλο κομισιόν της ιστορίας. Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, όχι μόνο στον αριθμό των θέσεων, αλλά και για τις πολιτικές που θα πρέπει να υλοποιούνται. Μια από αυτές θα έπρεπε να είναι να προσπαθήσουμε προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το, την πληγή της ε, ανδρικής βίας κατά των γυναικών. Επίσης, δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε τους πολίτες που έχουν ανησυχίες για το ότι ε, αδειάζουν οι περιφέρειές τους ε, λόγω της έλλειψης ευκαιριών. Θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης ε, με πόρους που θα βοηθήσουν στην οικολογική μετάβαση ώστε αυτή να είναι κοινωνικά δίκαιη και να μην αφήνει κανέναν πίσω. Έχουμε πέντε χρόνια μπροστά μας για να δείξουμε πως η πολιτική μπορεί να δώσει λύση, ότι η, η ισχύ τη ενώση και ότι η Ευρώπη έχει να πει πολλά σε έναν κόσμο που όλο ένα και περισσότερο ε, συντεράζει. Δεν θα πρέπει να Στου στους ε, ρήτορες του φόβου. Ε, ξέρουμε πως μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ισχυρή κομισιόν, μια κομισιόν τολμηρή που θα μπορέσει να δώσει νέο δυναμισμό για να ξεπεραστούν οι παλιές πολιτικές. Οι νέοι στόχοι απαιτούν νέες μορφές πολιτικής, μια πραγματικότητα που είναι όλο ένα και πιο περίπλοκη. Και καλύτερη μέρα για να ανανεώσουμε τις αρχές μας, για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα βιωσιμότητα του κοινωνικού μας μοντέλο και να εξασφαλίσουμε τη συνοχή των πολιτικών μας είναι ακριβώ η στόχη της βιώσιμης ε, ανάπτυξης, Agenda 2030. Και χαιρόμαστε που χάρη στο δικό μας αίτημα ε, δεχτήκατε ότι κάθε επίτροπος μεμονωμένα αλλά και όλοι συλλογικά θα είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτών των αρχών καθώς και την ένταξή τους στο Ευρωπαϊκό εξάμεινο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η νέα, το νέο πράσινο σύμφωνο είναι η προτεραιότητα Τη τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρουμε ότι ο Τίμερ μα θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Το κλίμα δεν μπορεί να περιμένει. Και για μα, πέρα από την πράσινη ατζέντα, θα είναι μια μια ατζέντα σάντουιτς πράσινη απ' έξω, κόκκινη από μέσα. Ε, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανανεώσει την κοινωνική της ψυχή, να ε, τοποθετήσει τους αγώνες ε, τους κοινωνικούς στην καρδιά. Και αυτό σημαίνει περίπλοκες πολιτικές. Στην προηγούμενη θητεία θέσαμε τις βάσεις για ένα κοινωνικό πυλώνα που τώρα πρέπει να αναπτυχθεί. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες έχουμε μια ολόκληρη σειρά από προτάσεις για να ενισχυθεί ο κοινωνικό, ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας, όπως και η οικονομική και φορολογική αρχιτεκτονική της Ένωση. Να είστε βεβαία ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτό. Και οι ίδιε αρχέ, ε, του σεβασμού στην ανθρώπινη εξωπρέπεια, την αλληλεγγύη και την δικαιοσύνη θα πρέπει να προσανατολίσουν επίση την εξωτερική μα πολιτική, την οποία πρέπει να πω ότι δεν μπορούσε να είναι σε καλύτερα χέρια. Τα χέρια του Τζουζέπ Μπορέλ που έχει το τεράστιο έργο να ε, επιβάλλει τις αρχές μας ε, και τα συμφέροντά μας. Η ειρήνη και πολυμερής ε, συνεργασία σε έναν κόσμο που διαρκώς συνταράσσεται από νέα προβλήματα. Έτσι, να μην χάσουμε την ομιμότητά μας και να είμαστε συνεπείς και να είμαστε και φιλόδοξοι με τον επόμενο προπολογισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Τα νέα μας σχέδια χρειάζονται περισσότερα χρήματα και γι' αυτό η ομάδα μας θα είναι πολύ απαιτητική με το επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες ε, θα δεν θεωρούμε πως έχει χαθεί ο αγώνας για την περισσότερη δημοκρατικοποίηση της Ευρώπης. Θέλουμε να θυμίσουμε το σύστημα του speech and candidate και να συζητήσουμε και πάλι για εθνικά ψηφοδέλτια, για, μάλλον για διεθνή ψηφοδέλτια, διακρατικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομείται καθημερινά και γι' αυτό και είναι και τόσο θαυμάσια. Έλεγε ο Πολανής Πακ, ένας από τους ε, πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα ε, επιστημονικά πειράματα αποτυχάνουν μια-δύο φορές πριν να επιτύχουν. Το, ε, δεν θα μπορεί να συμβεί κάτι ε, άλλο για την ευημερή μας ενωμένη και ισότιμη Ευρώπη. Σε αυτή τη θητεία θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στο, στο ε, όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες να ε, εμπιστευτούν ξανά τους θεσμούς. Εμείς οι σοσιαλιστές δημοκράτες είμαστε ξεκάθαροι. Ξέρω, θέλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και γι' αυτό σήμερα με την ψήφο μας, την απαιτητική, την πιστή και την άγρυπνη θα εμπιστευτούμε αυτό, ε, αυτή την Επιτροπή. θέλουμε η Κομισιό να το γνωρίζει και να ενεργήσει με υπευθυνότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τσόλος, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καρπός διαδικασίας σοβαρών εξετάσεων που έκανε το Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να ισχυροποιηθεί. Θα πρέπει τώρα να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι υποχρεώσει που ανέλαβε και που παρουσίασε η κυρία Βαντελάιν εδώ Ζητώ από αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δείξει τρία πράγματα, όραμα, πάθος και φιλοδοξία. Είναι ο μόνος τρόπος προετοιμασίας στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τα, τις νέες προκλήσεις του κόσμου και να ενθουσιάσει ταυτόχρονα τους λαούς. Χρειαζόμαστε ενθουσιασμό για να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα. Μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωπολιτική, είπε η κυρία Βαντελάεν. Πολύ καλό αλλά αυτό απαιτεί αλλαγές εις βάθος. Σαν ομάδα προωθήσαμε τρεις, τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες. Εν πρώτης, έχουμε τη φιλοδοξία η Ευρώπη να γίνει η πρώτη ήπειρος που θα είναι ουδέτερη σε άνθρακα το 2050, αλλά με μια οικονομία έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Αυτό θα είναι εφικτό με επιχειρηματίε με γεωργού και ερευνητέ που θα είναι έτοιμοι να δράσουν. Να επενδύσουμε λοιπόν στη μετάβαση με, μια, με ένα ταμείο δίκαιη μετάβαση και μια τράπεζα για το κλίμα και ένα προπολογισμό που είναι, ανταποκρίνεται στο ύψο των περιστάσεων. Δεύτερον, το ψηφιακό θέμα η ψηφιακή τεχνολογία μεταμορφώνει τι κοινωνίε μα με σημαντικέ ευκαιρίε που δημιουργούνται για του πολίτε, για την οικονομία μα, αλλά και με κινδύνους έναντι αυτών των εξελίξεων ας δημιουργήσουμε ηγετικέ εταιρείε σε αυτόν τον τομέα και α δώσουμε στις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις τη δυνατότητα πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κατάλληλο για την τεχνητή νοημοσύνη και πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για τα στοιχεία και τα δεδομένα. Είμαι σίγουρο ότι η Μαργαρέτε Βεστάγκερ και ο Μπρετών θα ανταποκριθούν στο ύψο των περιστάσεων. Ε, τρίτον, η Ευρώπη σε πέντε χρόνια θα μιλά ακόμα σε ισότιμη βάση με την Κίνα και τη ΣΥΠΑ. Θα είναι ακόμη μία φωνή που θα ακούεται στην Αφρική. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε μια πολιτική ασύλου και μετανάστευσης ανταποκρινόμενη στις αξίες μας και να οικοδομήσουμε μια εμπορική πολιτική έχοντας ρήτρες βιωσιμότητας που θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά και μια πραγματική Ευρώπη της άμυνας που θα είναι ανοιχτή όμως σε συνεργασίες. Και για όλα αυτά θα πρέπει να ξανασυνδέσουμε τους πολίτες με την Ευρώπη. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία που δεν θα καταλήγει σε εκλογές κάθε πέντε, θα επιλύονται τα προβλήματα μόνο κάθε πέντε χρόνια. Όλοι θα συμμετέχουν συνεχώς και η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αυτό το στόχο έχει όπου εκεί θα είναι κινητήρια δύναμη σε αυτό το συνέδριο ομάδα μου. Θα πρέπει τα θεσμικά εμπόδια να έρθουν, που εμποδίζουν ε, την Ευρώπη να κινηθεί όπως πρέπει. Το σύνδρομα του too little too late θα πρέπει να εκριζωθεί άπαξ